μια συζήτηση ε, και να τα συμφωνήσει, να τα βρει πριν ολοκληρωθούν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Οπότε δεν πειράζει, α πάμε και σε δεύτερη ανάγνωση αν χρειαστεί. Αλλά ελπίζω πάντω ότι αύριο θα συγκεντρώσω εντυπωσιακή πλειοψηφία για την έκθεσή μου. Εδώ τελειώνει η συζήτηση, λέει πρόεδρος, και θα ψηφίσουμε αύριο για την έκθεση του κυρίου Μάντερ. Next item on the agenda is report by Madame η επόμενη έκθεσή μα αφορά την κυρία Ρούλη. Την κυρία Ρούλη, μάλλον την έχει συντάξει και είναι οι νέε εξελίξει στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Και θα δώσω τώρα στην κυρία Ρούλη για τέσσερα λεπτά το λόγο. Παρακαλώ. Ελπίζω ότι τώρα με ακούτε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή συνεργασία που είχαμε και για το μέχρι του καλό αποτέλεσμα στην Επιτροπή. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εκθέσεώς μου. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους συμβαλωμένους ε, και αυτούς που αναθέτουν την εργασία και αυτούς που την αναλαμβάνουν και ε, κατακρίνουμε επίσης διότι υπάρχει μία περίπλοκη αλληλεπίδραση των νομοθεσιών που δεν μπόρεσε, να ανοίξει ε, την αγορά των δημοσίων συμβάσεων όπως ε, είχαμε προβλέψει το 2004 διότι χρειάζεται επίπονες και μακροχρόνιες διαδικασίες ε, είναι εις βάρος της ποιότητος αυτό και το αποδεικνύουν και οι μελέτες διότι τελικά αντί για την καλύτερη προσφορά επιλέγεται η πιο φτηνή ε, προσφορά και ε, δεν υπάρχει καμία μνήα για το δίκαιο εμπόριο ή για την καινοτομία. Είναι θέματα στα οποία η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί περαιτέρω. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πολλές αποφάσεις πρόσφατες έχει κατακρίνει την ασάφεια και έχει ζητήσει να υπάρχει μία ενίσχυση της εποπτείας, ιδίως όταν ε, πρόκειται για πολεοδομικά ε, ε, προγράμματα παραδείγματος χάρη αντί να περιλαμβάνεται μόνο ένα γενικό πλαίσιο εις, την, τα θέματα αυτά και τέλος παραμένουν οι εκχωρήσεις των δημοσίων οργανισμών παροχής υπηρεσιών όπου θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και να λάβουμε υπόψη τις ε, πολιτιστικές αλλαγές. Πράγμα το οποίο έχει ληφθεί υπόψη από όλους, είτε πρόκειται για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή τέλος και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, πράγμα το οποίο ήθελα να τονίσω στο έγγραφό μου. Ε, ένα τελευταίο θέμα είναι ότι οι δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσει οι δημοκρατικοί θεσμοί να χάσουν ε, το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας και γι' αυτό όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις ε, είτε για την αγορά καφέ ή άλλων προϊόντων είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τους θεσμούς και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η Επιτροπή να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και να τη συμβουλεύσει αντί να ξεκινά μία διαδικασία στην οποία παραπέμπει τις οργανώσεις αυτές για τα σφάλματα τους διότι δεν νομίζω ότι έτσι επιτυχάνει επιτάνεται ο στόχος τον οποίο επιζητούσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Βλέπω ότι τώρα υπάρχουν πολλοί ομιλητές οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο και σας υπενθυμίζω ότι κάθε ένας από εσά έχει ένα λεπτό. Ε, δίνω το λόγο καταρχήν στον κύριο Έγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να την ευχαριστήσω για την ουσιαστική εργασία την οποία έκανε και την διαθεσιμότητα την οποία επέδειξε για την συνεργασία μαζί μας για να καταρτιστεί η έκθεση αυτή η οποία προσπαθεί να βελτιώσει την νομική ασφάλεια διότι δεν θέλουμε να προτείνουμε περισσότερη νομοθεσία ηγεσία με κάθε κόστος αλλά να υπάρξει μεγαλύτερη προσβασιμότητα και μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Ένα βασικό θέμα το οποίο ανέφηξε η κυρία Ρούλε ε, είναι ότι ε, υπάρχει μία ευαισθησία και οδήγησε σε αντιπαράθεση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι εφόσον ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να μας προτείνει νέα στοιχεία νομοθετικά επί του θέματος αυτού θα την παρακαλούσαμε να ε, το πράξει λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς εφόσον υπάρχουν ε, νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες επί του θέματος. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Χωρίς μικρόφωνο. Α. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική μου ομάδα ε, θα είχε ε, υπερψηφίσει αυτή την έκθεση γιατί έχει πολλά θετικά στοιχεία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν τρία σημεία τα οποία δεν αναφέρονται και δεν μπορούμε να τα δεχτούμε όπως παρουσιάζονται. Καταρχήν ότι δεν ήταν δυνατόν να δεχθούμε από την κυρία Ρίλε ότι όντως υπάρχει ένα νομοθετικό πολιτικό ε, ε, πλαίσιο για τα οικονομικά συμφέρεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον τομέα των ε, κοινωνικών υπηρεσιών. Και ένα σημείο το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε καθόλου είναι αυτή η απόρριψη ε, ε, των αναθέσεων της παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτό δεν το δεχόμαστε, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό το έχει ρυθμίσει. Άρα δεν είναι πολιτική αντιμετώπιση. Πρέπει να πούμε σαφώς τι ζητάμε, εφόσον ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτήσει ένα ε, νομικό κείμενο το οποίο θέλει να μας υποβάλει. Πρέπει να πούμε σαφώς τι ζητούμε τι απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν της αποφάσεως της θετικής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δικαστηρίου κατά τρόπον ώστε να υπάρχει νομοθετική ασφάλεια και νομική ασφάλεια γι' αυτό και υποβάλαμε μία τροπολογία και καλούμε τους συναδέλφους να την υπερψηφίσουν. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ. Ο κύριος Μπουζόη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια προς την ε, ε, εισηγήτρια. Γιατί θα πρέπει όντως να έχουμε όσον αφορά τη δημόσια συμβάση περισσότερη διαφάνεια. Ε, έχουμε ήδη σε πάρα πολλές κρατασμένες πάρα πολλές προσφυγές και αυτό προέρχεται και από την πολυνομία. Αυτό ισχύει και για τη χώρα μου και δικονομικά προβλήματα έχουμε. Έχουμε επομένω προβληματική εφαρμογή του δικαίου. Ε, και η συνέπεια τελικά δεν μπορούμε να ωφεληθούμε από τα διευθυντικά ταμεία. Επομένω χρειαζόμαστε σαφέστερη καλύτερη νομοθεσία. Ε, αυτό θα μα διευκόλυνε πάρα πολύ. Κάτι άλλο τρόπο θέλω να σα πω αφορά το θέμα του, του κατωτάτου ε, ορίου. Όντω δεν θα πρέπει να γίνεται η επιλογή μόνο με αυτό το κρατήριο. Δεν πρέπει να γίνεται μια στάθμιση μεταξύ απόδοσης, αξίας και τιμής. <clears throat> Άρα, αφού να θεωρούμε αυτή την νομοθεσία, θα πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι και αυτό το κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Να καταλήξουμε σε κάποια ξεκάθαρα κριτήρια για να μην ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Να υπάρχει ασφάλεια του δικαίου και να αποφύγουμε διαφθορά. Ευχαριστούμε κύριε Χάρμπορ, ήρθε τώρα εσεί το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Όπω είπε ο σκιώδη τη πολιτική μου ομάδα, είμαι ο πρόεδρο τη ε, Νομικής Επιτροπής. Συγχαρητήρια προς την Χαϊντή Ρίλε γιατί είναι σημαντική η έκθεσή της. Κρίμα, κρίμα γιατί λόγω κάποιων παραδόξων διαδικαστικών μας διατάξεων μια τόσο σημαντική έκθεση για ένα τόσο σημαντικό θέμα της ενιαίας αγοράς και γενικά πολιτικής συζητείται με μονόλεπτες ομιλίες. Πάλι καλά που εδώ είναι ο κύριος Σταγιάννη. Γιατί? Θέλω να του πω ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ενθαρρύνουμε καινοτόμε επιχειρήσεις. Ο κ. Μπαρνία, βέβαια, θα ασχοληθεί και αυτός με το θέμα. Ελπίζουμε κάτι να κάνει και εκείνο. Όμως το θέμα είναι ότι, όπως λέει η έκθεση, αυτά που ισχύουν σήμερα φέρνουν σύγχυση. Είναι περίπλοκα. Και οι δημόσιες συμβάσεις γίνονται με ένα καθεστώς μάλλον τέτοιο έλλειψης ε, σαφήνειας. Αντί να είναι ένα εργαλείο, τόσο να δίνονται ευκαιρίες στην καινοτομία. Και έστω να φτάνουμε σε κάποια προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον και αντίστοιχε ε, υπηρεσίες. Άρα, πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτήν. Όλοι οι συναρμόδιοι επίτροποι να μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να διεκπαιρέσουμε αυτή την έκθεση. Πάσκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε κάτι με τις δημόσιες συμβάσεις. Πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος τους ώστε να έχουμε ε, ε, την εμπορία ή την αγορά κάποιων ε, εμπορευμάτων. Ε, θα πρέπει επίση με αυτή την νομοθεσία να καταφέρουμε να, διο... καταπολεμήσουμε την διαφθορά, να μπορούμε να έχουμε ένα απλουστευμένο νομοθέτημα και όλα αυτά να γίνονται μέσα σε συγκεκριμένε προθεσμίε. Άρα θα πρέπει να μπούμε ναι σε αυτή την έκθεση γιατί η εμπειρία μα έχει καταδείξει ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε την δέουσα ε, σύγκριση ε, θα πρέπει να έχουμε συμβάσεις που να είναι ξεκάθαρες και αυτές τελικά κερδίζουν το παιχνίδι ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο. Επίσης η εμπειρία μου έχει δείξει ότι πολλές φορές σε κάποιες ε, τοπικές, ε, σε κάποιους δήμους, κοινότητες, τοπικές αρχές έχουμε έγκριση συμβάσεων που πολλές φορές είναι ύποπτη. άρα καλύτερο να υπάρχει συγκρισιμότητα των, των, των συμβάσεων και αυτό μπορεί να βοηθήσει το διαδίκτυο. Έχετε το λόγο κυρία, το μικρόφωνο Θεωρώ ότι αυτή η έκθεση πέρασε, ξέρετε, στην Επιτροπή τη διασφορά με απόλυτη πλειοψηφία και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την Κομισιόν να αναθεωρήσει τη σχετική οδηγία. Αυτό που θέλουμε είναι οι δημόσιε συμβάσει να είναι πιο προσβάσιμε στι ΜΜΕ και έτσι οι διαγωνισμοί να είναι λιγότερο γραφειοκρατικοί, να επιδέχονται έλεγχο και εποπτεία. Βέβαια, ξέρετε εδώ πέρα, ε, το πρόβλημα είναι τι γίνεται του διασκευαστικό τομέα. Εκεί έχουμε πολλέ φορέ φαινόμενα διαφθορά. Πάντω, ε, δυστυχώ δεν θα προωθεί η δική μου τροπολογία. Ε, θα βοηθούσε η δική μου τροπολογία να να υπάρχει αυτή, αυτή η πύλη διαδικτυακή όπου θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει και να, να δει τα υπόπτα στοιχεία και, και, και άλλα χρήσιμα. Μόλι πάντω εκριζώσουμε τη διαφθορά, τότε οι ΜΜΕ θα θα μπορέσουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στι ε, δημόσιε συμβάσει και διαγωνισμού. Κύριε Τικάουτο, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. 16% του ΕΠ είναι ο τζίρος από αυτές τις δημόσιες συμβάσεις. Άρα αυτό που θα πρέπει να γίνεται είναι όλες οι ΜΜΕ να έχουν προσβασιμότητα. Αυτή η οδηγία παρέχει κάποιες εγγύσεις ούτως ώστε πάσα εταιρεία στην Ευρώπη να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της διαδικτυακά. Και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επίσης θα πρέπει να καλύπτεται από αυτή μας τη ρύθμιση ε, και να είναι δυνατόν να έχουμε και διαγωνισμούς με του διαδικτύου. Επομένω, θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό αυτή η πρόταση, αυτή η έκθεση. Ε, πάρα πολύ σωστές διατάξεις όσον αφορά τους ε, πιστωτές και πάρα πολύ θετικές διατάξεις για την ηλεκτρονική υπογραφή. Έχουν δεσμευτεί τα κρατημέλια όσον αφορά το 15% αυτών των διαγωνισμών ότι θα γίνεται με τρόπο ηλεκτρονικό. Η Ρουμανία, ξέρετε, ήδη έχει περάσει σχετικά μέτρα και νομίζω ότι έτσι έχουμε πετύχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη προσβασιμότητα από τα ΜΜΕ. Schwab. Ο κύριος Σουάμπ ζήτησε το λόγο και του τον δίνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε <clears throat> και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρούιλε σαν εισηγήτρια για αυτή την ε, πολύ καλή έκθεση διότι πρέπει να σας πω ότι το ΕΛΚ είναι ικανοποιημένο σε πολλά σημεία αυτής της εκθέσεως διότι έχουμε συμφωνήσει. Βέβαια δεν μπορεί κανείς ε, στο κοινοβούλιο αυτό να επιβάλλει τη δικιά του θέση αλλά νομίζω ότι μπορούμε έτσι να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία σειρά θεμάτων. Παραδείγματο χάρη, πώς είναι δυνατόν να δώσουμε κάτι ή στι αρχές κατά τρόπον ώστε ε, όταν υπάρχουν δημόσιε προμήθειε ε, να ε, οργανώνονται σεβόμενοι τις, τους κανόνες εσωτερικής, αγορά, εσωτερικής αγοράς. Πώς είναι δυνατόν να συνάδουν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται με την εσωτερική αγορά και πώς είναι δυνατόν να υπάρξει μία νομοθεσία η οποία θα αποβεί προς όφελος της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι στα σημεία αυτά έχουμε επιτύχει μία θετική πρόταση και ελπίζω ότι θα την υπερψηφίσουν και οι σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπασέσκο έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, βιώνουμε μια πολύ σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η κυβέρνησή μου αναγκάστηκε να μειώσει τους μισθούς στη Ρουμανία και να καταργήσει πολλές επιδοτήσεις. Αυτά ήταν πάρα πολύ σκληρά μέτρα γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε βέβαια ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται με διαφανή τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο και γι' αυτό πρέπει να βελτιωθούν και οι τρόποι με τους οποίους εξελίσσονται οι δημόσιες προμήθειες. Πρέπει έτσι να μειώσουμε τις απάτες, να μειώσουμε τη διαφθορά, γιατί υπάρχουσα γραφειοκρατική και περίπλοκη δομή της νομοθεσίας δεν μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον. Όλα αυτά ξέρετε ότι σε κάποιες ε, πολλές ε, αναθέσεις που θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει έχουμε οδηγηστεί σε πάγωμα των διαδικασιών και ε, μετά από νέες προσπάθειες θα ψηφίσουμε το νέο νόμο την 1η Ιουνίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η οικονομική κρίση έχουν υπογραμμίσει θα έλεγα τον σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζουν οι δημόσιες προμήθειες που θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους που είναι η ενθάρρυνση ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η τόνωση του ανταγωνισμού. Πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες και πρέπει να οδηγηθούμε σε μια περαιτέρω νομική βεβαιότητα με μεγάλη διαφάνεια ιδιαίτερα με ε, τα μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε στενότερη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας μας και πρέπει να προλαμβάνουμε τις διακρίσεις οι οποίες θίγουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχαίρω τους συναδέλφους και θα υποστηρίξω την πρόταση αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη, τελευταίος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο βρισκόμαστε ε, στη σημερινή κατάσταση την οικονομική στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι ο ρόλος τον οποίο έπαιξαν τα πιστοτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη ακεραιότητας και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα, δημιούργησε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι επανειλημμένα εξόδευαν πολύ περισσότερα από όσα είχαν και γι' αυτό λοιπόν τα μέτρα αυτά τα οποία θα βοηθήσουν την διαφάνεια είναι καλοδεχούμενα. Αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για τις προμήθειες αυτές θα πρέπει να έχουν την μέγιστη δυνατή επαϊοσύνη και να γνωρίζουν καλά και τις παράλληλες διαδικασίες. Πρέπει να υπάρξει απλούστευση βέβαια των διαδικασιών, δεν πρέπει να ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο και χρήματα για κάποιες διαδικασίες όταν δεν παρουσιάζουν προβλήματα επιπλέον. Ο κύριος Σταγιάννη να κλείσει τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Μπαρνιέ, τον οποίο αντικαθιστώ σήμερα, ακολούθησαν με πολύ μεγάλη προσοχή την προετοιμασία της έκθεσης πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για τις δημόσιες αγορές και προμήθειες. Μια σωστή πειθάρχηση, αν θέλετε, των διαδικασιών αυτών είναι σημαντικό πράγμα για να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις αυτές για το καλό των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είπαν οι προλαλήσαντες βουλευτές, ιδιαίτερα στο σημερινό πλαίσιο δημοσιονομικών πιέσεων οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της σχεδίασης των νέων τροπολογιών. Κάποιες από τις πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ξεκινήσει την εκτονιστέρων αναθεώρηση της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες. Έχουμε προσπαθήσει να διευκρινίσουμε τους κανόνες και για την αηφόρο ανάπτυξη και για την καταπολέμηση του αποκλεισμού. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, των αποφάσεων μάλλον του δικαστηρίου θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε το πεδίο συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα πλαίσια των δημοσίων προμηθειών. Σχετικά με μία πιθανή πρωτοβουλία λοιπόν για τις εκχωρήσεις, εμείς εδώ θα ακολουθήσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιπτώσεων που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και που είναι προϋπόθεση για η αδίποτε άλλη νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, από ό,τι φαίνεται το σημερινό νομικό πλαίσιο λειτουργεί ως τροχοπέδι τους της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει εφόσον κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή με μεγαλύτερη διαφάνεια και με μεγαλύτερη ε, θα έλεγα ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και γι' αυτό η αρχή της ανταπόδοσης είναι στη βάση ασδήποτε εμπορική συμφωνία την οποία συνάπτουμε. Και ζητούμε από το Κοινοβούλιο να διατηρήσει την ήδη δεδομένη σήμερα δεκτικότητα του και συμμετοχή του στη συζήτηση. Τέλειωσε η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Ρούιλε